Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους προσκεκλημένους μας. Ξεκινάμε το, το δεύτερο τμήμα της ε, συνεδρίασής μας, της Επιτροπής Ρέτζι. Το κύριο θέμα που έχουμε σήμερα το πρωί είναι ανταλλαγή απόψεων με τον Λετωνό ε, με την Λετωνική Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες για τα θέματα στα οποία είμαστε εμείς ε, αρμόδιοι. Πρόκειται για μια συμπληρωματική ανταλλαγή απόψεων προς την ανταλλαγή απόψεων που έγινε χθε με την κυρία Κρέτσου. Υπογραμμίζεται η σημασία της πολιτικής συνοχής και στην, στην μείωση των ε, κοινωνικών ανδικιών και την ε, καταπολέμηση της ε, ανεργίας για να διασφαλιστεί ότι θα ξεκινήσει ομαλά η νέα προγραμματική περίοδος. Η νέα Προεδρία θα δώσει σημαντική ε, προσοχή στην αναθεώρηση της πολιτικής για την περιφερειακή συνοχή, την αστική ατζέντα και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Από την πλευρά μου καλωσορίζω και χαιρετίζω τις απόψεις ε, του Υπουργού για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στις θέσεις απασχόλησης στην, στην πολιτική συνοχής. Προτείνω να ακολουθήσουμε την ε, συνήθη διαδικασία για την ανταλλαγή απόψεων. Θα καλέσω πρώτα τον Υπουργό να μας παρουσιάσει τις θέσεις του και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής για να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, ξεκινώντας με τον κύκλο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν δίνω τώρα το λόγο στον Υπουργό Οικονομικών ε, στον εκπρόσωπο της Προεδρίας, της Λετωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου, τον κύριο Γιάννη Ρέσο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή που, μου, που διοργάνωσε χθες η Πρόεδρος. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω κάποια από τα μέλη της Επιτροπής. Και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε την ε, πολιτική συνοχή που είναι από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση και την ανάπτυξη. Φέτος είναι η 25η επέτειος ανεξαρτησίας της Λετωνία από το ολοκληρωτικό καθεστώς τη Σοβιετική Ένωσης. Δέκα χρόνια από την προσχώρηση τη Λετωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα χρόνο από τότε που προσχώρησε στην Ευρωζώνη. Το να αναλαμβάνουμε την ε, Προεδρία του Συμβουλίου είναι και μεγάλη μας τιμή και μεγάλη ευθύνη για μας. Η Λετωνία θα αξιοποιήσει την Προεδρία για να ακολουθηθούν, να, ε, ε, να υπηρετηθούν οι πολιτικές και να αντιμετωπιστεί η κρίση. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα βελτιώνουν την καθημερινή του ζωή. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους, τα θεσμικά όργανα επιτέλεσαν μεγάλο ε, πολύ έργο για ε, να θεθούν οι προτεραιότητες για τη νέα περίοδο. Αυτές οι προτεραιότητες καθορίστηκαν στο πρόγραμμα της, ε, του Τρίου της Προεδρίας, της Κομισιόν και στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2015. Η Λετωνική Προεδρία έχει καθορίσει τρεις προτεραιότητες. Ανταγωνιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφιακή Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολιτική της συνοχής είναι ε, μία από τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας, συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα, και με το όραμα της νέας Επιτροπής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και το πρόγραμμα εργασιών για το 2015. Θέλουμε να συνεχίσουμε να, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, βρίσκονται... ε, ε υλοποιούνται αυτή τη στιγμή από, τη, από τις χώρες. Η, η ανάπτυξη μπορεί να φέρει νέες θέσεις απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα παίξει κρίσιμο ρόλο η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής που θα βασίζεται σε τρία στοιχεία. Προτού σας παρουσιάσω λεπτομερώς τις προτεραιότητες Προεδρίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας μεταφέρω την λεπτονική εμπειρία. Η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας μου. Έχει δημιουργήσει την, τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη συμμετοχή της Λετωνίας στην εσωτερική αγορά και μα έδωσε την ευκαιρία ε, να προσχωρήσουμε στην Ευρωζώνη. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΑΕΠ κατά κεφαλή ήταν μόνο 47% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2013 όμως είχε ήδη ανεβεί στο 67% το ποσοστό αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι παρά την κρίση, στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών η Λετωνία έχει ε, προσεγγίσει το βιωτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 20%. Πρόκειται για μεγάλο επίτευγμα και σημαντικό ρόλο έπαιξε η συγχρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και τέτοιου, τέτοια, είδους εξέλιξη υπάρχει και στις τρεις βαλτικές χώρες αλλά και στις περισσότερες νέες ε, χώρες. Η κρίση έπληξε την, κρίση, την Λετωνία ε, με, πολύ έντονο τρόπο. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% και έτσι τα, η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία ήταν ζωτική σημασία. Προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν ε, να ε, εφαρμοστούν τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια επενδύσεων. Το πρόγραμμα επενδύσεων αξιοποιήθηκε για, να, για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών. Συνολικά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανήλθαν σε 70% των δημόσιων επενδύσεων. Χθες συζητήσαμε για τα ταμεία και διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό στη Βουλγαρία είναι παρόμοιο. 73%. Το 2011 επήλθε η ανάκαμψη στη Λετωνία λόγω της ε, στιβαρής δημοσιονομικής πολιτικής και της βοήθειας από τα ε, ευρωπαϊκά ταμεία και έτσι καταφέραμε να ζήσουμε μια αναγέννηση βασισμένη στις εξαγωγές. Η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είναι από, τα υψηλό, από τις υψηλότερες ε, που έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια, 1,8 σε 2,1%. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πολιτική. Και στις προηγούμενες περίοδους είχαμε διαρθρωτικά προβλήματα στην παιδεία, την απασχόληση, την, ε, τις μεταφορές, για να αναφέρω μερικά παραδείγματα μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει πολύ σημαντικά στις δημόσιες επενδύσεις στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο η τα αποτελέσματα της πολιτικής έχουν ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κυβέρνηση, τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα προβλήματα της Λετωνίας είναι η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλή κοινοτομία, φτώχεια και ανεργία. Αυτές είναι οι προκλήσεις που θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε, να αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Ταμείων την περίοδο 2014-2020. Θα συνεχίσω τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να αποτελέσει η πολιτική συνοχή σημαντικό πυλώνα της πολιτικής στη Λετωνία. Ξεκινούμε λοιπόν την Προεδρία στην, στην αρχή αυτή τη νέα επενδυτική περίοδου 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικέ οικονομικέ προκλήσει, χαμηλή ανάπτυξη, ψηλή ανεργία, χαμηλό επίπεδο επενδύσεων. Η αναθεωρημένη κοινων, ε, πολιτική συνοχή είναι ένα από του πυλώνες που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Χρειάζεται, χρειάζονται προσπάθειε από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη για να επιταχυνθεί το πρόγραμμα υλοποίησης. Το οποίο ωστόσο αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει εγκριθεί. Τον Δεκέμβριο το Συμβούλιο υποστήριξε το επενδυτικό ε, σχέδιο του κυρίου Γιούγκερ, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Παρομοίως, η ανακοίνωση Κομισιόν καλεί στην ε, επέκταση των, ε, της χρήσης των ταμείων αυτών στην ε, χάραξη των πολιτικών. Επιπλέον, στα τέλη της τελευταίας χρονιάς, το ζήτημα της πλήρους αξιοποίησης των ταμείων την προηγούμενη περίοδο τονίστηκε. Η Κομισιόν εργάζεται δραστήρια με τα κράτη-μέλη για να αξιοποιηθούν για να αξιολογηθεί η χρήση των, ε, των ε, ταμείων, των κοντιλίων την προηγούμενη περίοδο. Το δεύτερο εξάμεινο του 2014 η Κομισιόν ε, διοργάνωσε συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Αστική Πολιτική προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το αν χρειάζεται και αν και κατά πόσο χρειάζεται μια τέτοια πολιτική. Λαμβάνοντα υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και τα επιτεύγματα τη Ιταλική Προεδρία, θα συνεχίσουμε το έργο στο Συμβούλιο. Μία από τι προτεραιότητέ μα θα είναι να καταλήξουμε στη συμφωνία για τι τροποποιήσει του ε, πολιετού δημοσιονομικού πλησίου που χρειάζονται για να βελτιωθούν τα ε, τα προγράμματα που προβλέπονται για την περίοδο 2014-2020. Το, η Λετωνική Προεδρία προσβλέπει προς την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα. Μια από τις προτεραιότητες μας είναι το επενδυτικό σχέδιο το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε καλό προγραμματισμό στην αρχή της περίοδου, κάτι που θα μας ε, επιτρέψει ε, την ε, ενδεδειγμένη αξιοποίηση των κονδυλίων. Επιπλέον, χρειαζόμαστε διοικητικές ικανότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την αναθεωρημένη πολιτική και να καταλήξουμε στα στους στόχους που έχουμε θέσει. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι περιμένουν αποτελέσματα από αυτή τη νέα αναθεωρημένη πολιτική και μπορούμε να, να επιτύχουμε τα αποτελέσματα αυτά μόνο αν δημιουργήσουμε την πρακτική βάση για την εφαρμογή. Επίσης, θέλουμε να επεκτείνουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που έχει τύχει πλέον της υποστήριξης του Συμβουλίου κάτι που τονίστηκε και στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου, αυτό το Ταμείο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ταμείο που μπορεί να ε, συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πραγματικά μπορεί να προωθήσει τις επενδύσεις στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο πολύ πιο συντονισμένο. Η Λετωνική Προεδρία θα βασιστεί επίσης στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Ιταλικής Προεδρίας, σύμφωνα με τα οποία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν προγράμματα σύμφωνα με τις εθνικές συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να αξιολογήσουν βέβαια και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που τους δίνονται από τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται τον Ιούνιο μία συζήτηση για τα ζήτηματα αυτά σε μία άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Υπεύθυνων για την Πολιτική Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με τον της Περιφέρειας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, θα διοργανώσουμε μια συνδιάσκεψη για τις προκλήσεις που αφορούν τις περιφέρειες στην περίοδο 2014-2020. Στόχος της συνδιάσκεψης αυτής είναι να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ερευνητών και επιστημών από τη μία πλευρά και των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής από την άλλη. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική που θα βασίζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Κυρίες και κύριοι, η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής δεν αποτελεί μόνο ένα στρατηγικό μέσο ανάπτυξης και επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά προβλέπει επίσης και πάρα πολύ σημαντικά μέσα για την προώθηση της ε, περιφερειακής ε, συνοχής. Θα δώσουμε λοιπόν εμείς ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της ε, προώθησης της λεγόμενης Urban Agenda, δηλαδή των προτεραιοτήτων που έχουμε στον τομέα των πόλεων και της αστικής ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε στον τομέα αυτό την εργασία που ήδη έχουν ξεκινήσει οι προηγούμενες προεδρίες θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόθεση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον. Επίσης, περιμένουμε και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αστική αυτή διάσταση της πολιτική συνοχής και προσβλέπουμε σε πολύ θετικές επικοδομητικές συζητήσεις μαζί σας για το ζήτημα αυτό. Επίσης, από πλευράς Προεδρίας προωθούμε μία συζήτηση για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την εδαφική ανάπτυξη, ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει παρακώς μέχρι σήμερα. Το ζήτημα λοιπόν αυτό θα συζητηθεί στην σε άτυπο διακυβερνητικό επίπεδο. Το πιο, η πιο σημαντική, αν θέλετε, εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου άτυπη διάσκεψη των Υπουργών, η οποία είναι αρμόδιοι για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αστική ανάπτυξη, όπου θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε όλα τα ζητήματα εκείνα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων αλλά και των λεγόμενων μικρομεσαίων πόλεων και πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν στο γενικότερο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται επίσης και μία περαιτέρω απόφαση η οποία θα ληφθεί στα πλαίσια της παγκόσμιας διάσκεψης Habitat 3 το 2016. Βέβαια του στήματος αυτού θα επιληφθεί περαιτέρω η Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω η δική σα Επιτροπή περιφερειακή ανάπτυξη έχει συμβάλει πάρα πολύ σημαντικά στη διαμόρφωση τη νέα περιφερειακή πολιτική και τη πολιτική συνοχή για την περίοδο 2014-2020. Πραγματικά η πολιτική αυτή θα είναι πλέον μια επενδυτική πολιτική που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά προκειμένου αυτή η νέα πολιτική συνοχή να στεφτεί με επιτυχία, να εφαρμοστεί επιτυχώ στις περιφέρειες και πραγματικά να βελτιώσει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική συνεργασία με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω με την Επιτροπή σα Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στι ε, ερωτήσει σα όσον αφορά τι προτεραιότητε αυτέ τη Λετωνική Προεδρία. Προσβλέπω σε μια ειλικρινή και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτή την πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Τώρα θα δεχθούμε τις ερωτήσεις του ακροατηρίου. Ξεκινούμε με τις ερωτήσεις των συντονιστών. Ο κύριος Φανίστερο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Ως προς την παρουσίασή σας, κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για επενδύσεις Μιλήσατε για το ότι θέλετε να κάνετε τα πράγματα σωστά. Μιλήσατε για πόλεις, για δήμους, για κοινότητες, για περιφέρειες. Όλα αυτά να γίνουν πιο ορατά στον Ευρωπαίο πολίτη. Ως προς τα επιτεύγματα της Ιταλικής Προεδρίας, από ό,τι φαίνεται, θέλετε να τα συνεχίσετε και να βασιστείτε σε αυτές τις επιτυχίες. Γιατί έξι μήνες βεβαίως δεν είναι αρκετοί. Σε κάθε περίπτωση, στα συμπεράσματα της Ιταλικής Προεδρίας λέγεται ότι η Λετωνική Προεδρία θα συνεχίσει με, στο δρόμο της Ιταλικής Προεδρίας. Δηλαδή, για να υπάρχει διάλογος τακτός στο άτυπο Συμβούλιο και όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και εξωτερικών υποθέσεων. Οι Ιταλοί έκαναν μία πρώτη συζήτηση για τη διακυβέρνηση, για την διοίκηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2020. Και τα υπογράμμισαν όλα αυτά και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η μεθοδολογία αυτή. Τους τελευταίους μήνες αυτό το έχουμε προσπαθήσει να το πετύχουμε, όμως ε, δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Ως προς τις προτεραιότητες τα Συμβούλια Υπουργών, το σημαντικό είναι να τονίσουμε τη συνοχή, όπως το είπατε και πολύ σωστά. Ε, και αυτό ήταν ε, προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας. Το σχέδιο επενδύσεων, το επενδυτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ είναι καλό κατά τη γνώμη μου. Με ικανοποιεί η παρουσίαση αυτού του σχεδίου, όμως δεν θα πρέπει να, ξεχνούμε, να ξεχνάμε ε, πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις. Μιλούμε για 460 δις ευρώ και πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη. Με το σχέδιο Juncker μπορεί κανείς να πετύχει πολλά πράγματα το Συμβούλιο Υπουργών όταν θα ασχοληθεί με το θέμα της συνοχής, ε, το σημαντικό είναι να υιοθετήσει ξεκάθαρη επιτέλους θέση. Επομένως, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, ποια είναι η άποψή σας. Είστε διατεθειμένος να εμπλέξετε όλους στη συζήτηση αυτή. Τέλος, χθες ε, μιλήσαμε για τις μακροπεριφέρειες. Είπατε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η άποψή σας για τις μακροπεριφέρειες. Καλό είναι να μιλούμε για μακροπεριφέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει Όπως μιλούμε και για τη διεύρυνση, ε, καλό είναι να μην μένουμε στη θεωρία και στα πολλά λόγια. Έχουμε μακροπεριφέρειες, ας μην ε, πάμε πιο πέρα. Φτάνουν αυτά που έχουμε. Παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φανίλ Σεντρόιδη, κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι εκτιμάται ιδιαίτερα την πολιτική συνοχή και για τη χώρα σα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάλαβα ότι από την εμπειρία σας ε, η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους πυλώνες της επενδυτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε σχέση με το επενδυτικό πακέτο Juncker να Δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, πολιτική συνοχή και συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι το ερώτημα το ότι χρειαζόμαστε ένα συμβούλιο που θα ασχολείται με την πολιτική συνοχή. Ξεκίνησε μια τέτοια προσπάθεια από την Ιταλική Προεδρία και ορθώς. Εδώ και πολλά χρόνια το Κοινοβούλιο ζητά να υπάρξει, να θεσπιστεί Συμβούλιο Υπουργών για την πολιτική συνοχή. Δυστυχώς δεν ήμασταν ιδιαίτερη επιτυχής μέχρι τώρα και γι' αυτό τον λόγο υποστηρίξαμε με όλες μας τις ε, δυνάμεις την Ιταλική Προεδρία ως προς αυτό και από την ε, δική μας πλευρά, εκ μέρους της δικής μας ομάδας, θα ήθελα να σας καλέσω να συνεχίσετε την ε, δουλειά αυτή γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το επενδυτικό πακέτο να συνδυαστεί με την πολιτική συνοχής και νομίζω ότι το ζήτημα των επενδύσεων και της εξέβρεσης νέων πόρων δεν ε, ε, εξελίχθηκε με τον επιθυμητό τρόπο μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Όσον αφορά την αστική πολιτική θέμα που έχει θέσει στο πρόγραμμα εργασιών της και η Κομισιόν. Νομίζω ότι εν ώψη της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες στο συγκεκριμένο τομέα. Έχετε εσείς ε, εικόνα για το ποιες θα είναι οι προσπάθειες που θα αναλάβει η δική σας Προεδρία. Η χάρτα της λειψείας ε, έχει αρκετά χρόνια από τότε που ε, συμφωνήθηκε. Βρισκόμαστε βεβαίως στην, ε, στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης, υπάρχουν πολλά κοινωνικά προβλήματα και από αυτή την άποψη ενδεχομένως να χρειάζεται και μια αναθεώρηση της αστικής πολιτικής. Ποια είναι λοιπόν, ποιες είναι λοιπόν ε, οι δικές σας προσπάθειες για την προώθηση της, του συγκεκριμένου θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω το ECR να θέλει το λόγο. Κύριε Γιάκουφτσιτς, έχετε το λόγο. Э, Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό που ήρθε εδώ ε, και για την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε. Ε, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και εγώ πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα ζήτημα πραγματικά κεντρικό, ζωτικό για τη δική μας Επιτροπή και ευχαριστώ τον Υπουργό που επιθυμεί να συνεχίσει την πολιτική αυτή. Σίγουρα με βάση τη δική σας εμπειρία θα το πράξετε, αλλά θα λάβετε υπόψη και την άποψη των άλλων χωρών μελών και γι' αυτό θεωρείτε ότι η κατάσταση ε, των χωρών θα ήταν πολύ χειρότερη αν δεν είχαμε την πολιτική συνοχή. Είναι κάτι που εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε πολύ καλά. Χρειάζεται συνέργεια λοιπόν μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του σχεδίου Juncker. Πρέπει να λειτουργήσουμε έξυπνα και να έχουμε μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των παλαιών και των νέων ε, χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ των διαφόρων μέσων που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να μην αμφισβητήσει κανείς τα μέτρα, ε, τα επενδυτικά, τα οποία θα έχουν τεράστια σημασία τα επόμενα χρόνια. Είμαι πεπισμένος ότι εάν δεν καταφέρουμε να ε, πυροδοτήσουμε, να αναζωογονήσουμε ξανά ε, την ευρωπαϊκή οικονομία και μάλιστα στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, δεν θα έχουμε καμία αξιοπιστία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και σίγουρα θα θεωρηθούμε υπόλογοι και υπεύθυνοι για αυτό το οποίο θα έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Αυτό καταρχάς, κατά δεύτερο λόγο, η στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες. Σήμερα έχουμε τέσσερις, τη Βαλτική, το Δούναβη, την Αδριατική με τις Ιόνιους νήσους και τις Άλπεις. Τέσσερις μακροπεριφέρειες. Εγώ ανέκαθεν ήμουν υπέρ ε, της στρατηγικής για τις μακροπεριφέρειες. Πρέπει όμως να εξετάσουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής. Εκτός από τη Βαλτική και εν μέρη, εκτός και από το Δούναβι, η μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίων Νήσων μόλις τώρα συγκροτήθηκε Άρα δεν θα πρέπει να ε, κουράσουμε αν θέλετε αυτή την έννοια η οποία είναι καλή αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού στην Ευρώπη η έννοια της ε, μακροπεριφέρειας μην υπονομεύσουμε λοιπόν ε, το πρόγραμμα αυτό προτού καν αρχίσει ευχαριστώ η Πρόεδρος κυρία Βάνα έχετε το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλύσαντες, να τονίσω και εγώ πόσο σημαντική είναι για μας η αστική πολιτική, ιδιαίτερα για τους στόχους, ε, για την επίτευξη των στόχων για το 2020, η πόλεις έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και γι' αυτό το λόγο μας ενδιαφέρει ε, σας, ε, ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις, πώς θα ενισχύσετε τις πόλεις και από άποψη πραγματοποίηση επενδύσεων. Θα ήθελα όμως και εγώ να μιλήσω για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και συγκεκριμένα για το Δούναβι. Εγώ προέρχομαι από την Αυστρία και φαίνονται ότι υπάρχουν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ε, συντονισμού για αυτήν την ε, ε, μακροπεριφέρεια. Πρόκειται δηλαδή να δημιουργηθεί ένα νέο κέντρο συντονισμού, κάτι που και μάλιστα αυτός ο ε, μηχανισμός θα υποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ε, διακηρυγμένη πολιτική ε, που ήταν πάντοτε ε, ότι οι μακροπεριφέρειες οι ίδιες θα πρέπει να αποφασίζουν και να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Οπότε ποιες είναι οι δικές σας πολιτικές. Η κυρία Νταμάτο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για αυτό το σχέδιο Juncker το οποίο τόσο πολύ χαροποίηση ορισμένους, αλλά θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να διασκεδάσετε όλες αυτές τις ανησυχίες που πάρα πολλές πολιτικές ομάδες έχουν εκφράσει. Δεν καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στους στόχους της πολιτικής συνοχής και το συγκεκριμένο σχέδιο Juncker. Υπάρχουν επικαλύψεις υπάρχουν ε, αντιφάσεις, μπορούμε να καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτές τις δύο πολιτικές. Μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι υπάρχουν βέβαια όλα αυτά τα χέγγια στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αυτό ήταν ο πρώτος ε, γύρος ερωτήσεων και παρατηρήσεων. Να ζητήσω λοιπόν από τον Υπουργό να απαντήσει πρώτα σε ερωτήσεις αυτές και θα συνεχίσουμε με δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έχετε το λόγο. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τις προτεραιότητες καταρχάς και όσον αφορά την πολιτική συνοχής και πώς μπορεί αυτή να ενταχθεί, να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας. Ήδη εξ αρχής θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για όλη τη νέα περίοδο προγραμματισμού και ήδη στα τέλη του έτους θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδότησης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει όμως μια συζήτηση για την διοικητική ικανότητα, τη διοικητική υποδομή, που αποτελεί σημαντικότατη προϋπόθεση για την εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής συνοχής. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Επίσης, είναι θεμελιώδες να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα χρησιμοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό και ευφύ. Αυτό περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το σύστημα υλοποίησης των ε, χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ως προς αυτό το Συμβούλιο υποστηρίζει την ε, διοργανική υποστήριξη που ε, υπάρχει και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι αναγκαστικά μια πολιτική συνοχή υπαριθμών 2, αλλά θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έρθει να συμπληρώσει και να υποστηρίξει τα προγράμματα. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων αναφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τι προτιθέμεθα εμεί να κάνουμε ω προ αυτό. Καταρχά να σα πω ότι προφανώς εκτιμούμε και χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του σχετικού κανονισμού, ανακοινώθηκε εγκαίρος και προσβλέπουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε επεξεργασία της πρώτης αυτής κανονισμού στο Συμβούλιο. Έχουμε μάλιστα ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση αυτή κανονισμού όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα περάσει όσο δυνατόν πιο ανώδυνα και γρήγορα μέσα από τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τηρήσουμε αυτό το πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και να εγκριθεί εν γέρος ο νέος αυτός καονισμός. Προσβλέπουμε λοιπόν σε επικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Αυτό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το σχετικό σχέδιο επενδύσεων πραγματικά θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα οδηγήσει σε απτές επενδύσεις. Τώρα πώς συνδέεται με την πολιτική συνοχή και με τα διαρθρωτικά ταμεία. Καταρχάς, πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και θα δοθούν τότε και πιο συγκεκριμένε απαντήσεις. Και μόνο τότε εγώ θα μπορώ να σας δώσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία αφού έχει γίνει πρώτη συζήτηση σε επίπεδο ECOFIN. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Όσον αφορά τον, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το πώς συνδέεται μετά όσα συζητάμε. Η πολιτική συνοχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, όπως το είπαμε ήδη. Χαιρετίζουμε λοιπόν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων επί Ιταλικής Προεδρίας όσον αφορά την έκτη έκθεση πολιτικής συνοχής που πραγματικά καταδεικνύει και τη δράση που πρέπει να λάβουμε σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να έχουμε μια ρεαλιστική συζήτηση με τους υπουργού για όλα τα ζητήματα πολιτικής συνοχής προκειμένου οι συζητήσεις αυτές πραγματικά να οδηγήσουν σε προστιθέμενη αξία και αυτά αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα την πολιτική συνοχή και αν θα πρέπει αυτή να ενταχθεί στα πλαίσια των συζητήσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, εμείς είμαστε δεκτικοί ως προς την πρόταση αυτή θεωρούμε ότι όντως θα πρέπει στο Συμβούλιο αυτό να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία θα ενδυναμώσουν την πολιτική συνοχή και που θα ενισχύσουν επίσης την υλοποίηση του προγράμματος, των προγραμμάτων μάλλον που εντάσσονται στην περίοδο 2014-2020. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής ανταποκρίνονται όντως στις ελπίδες και στις προσδοκίες των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Eh, Το επόμενο ερώτημα για τις μακροπεριφέρειες και τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος αυτών των περιφερειών είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά την ε, συνοχή, την πολιτική συνοχή και θα μας επιτρέψουν τη χρήση των ε, υφιστάμενων δομών και εργαλείων χωρίς να δημιουργήσουμε ή να θεσπίσουμε νέους νόμους. Κατά τη γνώμη μας, οι μακροπεριφέρειες σχετίζονται με το να εξευρεθούν περισσότερα χρήματα, αλλά με την καλύτερη αξιοποίηση των ε, υφιστάμενων κονδυλίων. Και σε αυτό το τομέα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ιταλική Προεδρία για το γεγονός ότι προώθησε ε, την ε, δημιουργία της νέας μακροπεριφέρειας ε, Αδριατικής, Αδριατικής Ιουνίου. Περιμένουμε η Κομισιόν να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσεων για την τέταρτη μακροπεριφέρεια των Άλπαιων. Έχουν, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν και σε συνεργασία με την Κομισιόν θα ε, διοργανώσουμε το έκτο ετήσιο φόρουμ αναθεώρησης τον Ιούνιο για την αναθεώρηση της ε, μακροπεριφερικής στρατηγικής στην Βαλτική. Σε ό,τι αφορά την αστική πολιτική και το αστικό θεματολόγιο που ανέφεραν οι εκπρόσωποι των ομάδων, πρέπει να σας ομολογήσω ότι σε διάφορες συζητήσεις, σε διάφορα φόρα, σε διάφορα βήματα, έχει εκφραστεί η άποψη για προώθηση της αστικής πολιτικής, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συνένεση για το ποια θα πρέπει να είναι η μορφή αυτής της αστικής πολιτικής. Σίγουρα θα ε, ε, περιλαμβάνει την σύγκληση. Θα υπάρχει το πρόγραμμα αστικής ε, ανάπτυξης. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές, οι πόλεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αναλυθεί διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της αστικής πολιτικής, αλλά αυτή τη στιγμή οι πρωτοβουλίες αυτές δεν συγκλίνουν αυτό που πρέπει εμεί να διασφαλίσουμε είναι ε, η αστική πολιτική να είναι πιο στοχευμένη. Και σε τελική ανάλυση η αστική πολιτική δεν μπορεί να διακρίνεται, ε, να διαφέρει μάλλον από την ε, περιφερειακή πολιτική. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών ε, πόλεων. Πολλοί ενδιαφερόμενοι πιστεύουν ότι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ότι τα, προγράμματα ανάπτυξης θα πρέπει να δημιουργηθούν από τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Κομισιόν και τις ίδιες τις πόλεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες ε, δράσεις εκ θα πρέπει αυτές να ε, συντονιστούν ώστε να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Η δική μας Προεδρία έχει στόχο να αρχίσει τις συζητήσεις και να υπάρξει συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δημιουργία ενός προγράμματος αστικής πολιτικής που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των πόλεων και θα συμβάλλει στην ε, εδαφική ε, ανάπτυξη, στην ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις λοιπόν και η αστική πολιτική είναι μία από αυτές τις διαστάσεις που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Συνεχίζουμε με τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Μπόγκοβιτς είναι ο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας, να σας συγχαρώ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, για τα επιτεύγματα της χώρας σας τα τελευταία χρόνια. Έχετε υιοθετήσει τις μεταρρυθμίσεις, έχετε καταφέρει ε, να έχετε δημοσιονομική σταθερότητα και όπως είπατε και εσείς ο ίδιος στην αρχή, με την πολιτική συνοχής κατάφερε η χώρα σας να πλοηγηθεί σε πιο ήρεμα νερά παρά την οικονομική κρίση σήμερα. Στηρίζουμε τις θέσεις σας. Εμεί, εγώ είμαι από τη Σλοβενία. Δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις τόσο καλά όσο εσείς και δεν καταφέραμε να επιτύχουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα τόσο καλά όσο εσείς. Και γι' αυτό η κρίση παρατάθηκε στη Σλοβενία. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει ό,τι και εσείς εμείς εδώ στη Σλοβενία. Αυξήσατε το ΑΕΠ σας και ήσασταν στο 47% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είστε στο 67% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια τεράστια αύξηση αυτή. Στη Σλοβενία έχουμε φτάσει στο 85% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να το κάνουμε αυτό, πολύ περισσότερο από ό,τι σε εσά. Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί να, ε, της ομάδας που θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις που ε, παρουσιάζει η πολιτική συνοχή στο μέλλον. Αυτό χρειαζόμαστε για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί ανταγωνιστικότητα είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Τρίτη σας στόχος, τρίτη σας προτεραιότητα, η δράση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικό. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις ως προς το σχέδιο Juncker. Θα πρέπει να δράσουμε με σοφροσύνη, να υπάρχει σωστή αλληλεπίδραση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του σχεδίου Juncker για να έχουμε καλύτερη πρόοδο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σχέδιο Juncker για να αναζωπηρώσουμε την οικονομία σε όλες τις χώρες. Σήμερα έχουμε την τάση να ζούμε όλο και περισσότερο σε μεγάλες πόλεις αυτό προσφέρει πλεονεκτήματα, αλλά δημιουργούνται και προβλήματα. υπάρχει θέμα με την κινητικότητα, με την ποιότητα του αέρα, με τη δημιουργία θέσεις, θέσεων απασχόλησης, με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων μεταξύ άλλων. Και στο παρελθόν, ξέρετε, δεν είχαμε δώσει μεγάλη σημασία σε ένα από τα βασικά προβλήματα που είναι η ασφάλεια και η κοινωνική ένταξη, η ενσωμάτωση. Οι τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας τον τελευταίο μήνα αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι πάρα πολλά προβλήματα δημιουργούνται όλο και περισσότερο στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις λόγω της ανεργίας, λόγω του γεγονότος ότι ε, υπάρχουν αποκλεισμένοι, υπάρχουν περιθωροποιημένοι στις κοινωνίες μας, δυστυχώς, εξού και συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά την υλοποίηση των πολιτικών για το άστι δεν πρέπει να λησμονούμε το θέμα, το σκέλος της ασφάλειας. Ε, δεν λέω ότι μπορούμε να το λύσουμε αναπτύσσοντας τον στρατό. Αντιθέτως, εάν αναπτύξουμε σωστά τις πόλεις θα λύσουμε το θέμα της ασφάλειας. Ποια είναι η άποψή σας, πώς ε, πρέπει να δράσουμε σε, σε θέματα ασφάλειας και πόλεων. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ να συζητήσετε μαζί σας. Έχετε μιλήσει για το σχέδιο Γιούγκερ, Έχω όμως ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Μιλήσατε για ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα από τη μία και από την άλλη το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ρέτζι δείχνουν και τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να εμπλακούν οι περιφερειακές διοικητικές αρχές κατά την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου. Άλλωστε, τα δύο τρίτα των επενδύσεων στην Ευρώπη γίνονται από τις περιφερειακές αρχές. Επομένως, εάν εμπλακούν οι θύνοντες στο σχεδιασμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το συγκεκριμένο ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Εσείς και η Λετωνική Προεδρία, τι θα κάνετε κάνετε για να κινητοποιήσετε τα κράτη-μέλη να μην υποβάλλουν μόνο σχέδια το καθένα για τον εαυτό του, αλλά να εμπλέξουν και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην κατάρτιση των σχεδίων αυτών. Γιατί αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εμείς ευχαριστούμε. Επόμενο ερώτημα από τον κύριο Ρούλς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Καλώς ήρθατε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στη Λετωνική Προεδρία. Οι περισσότερες ερωτήσεις που ήθελα να θέσω έχουν ήδη τεθεί. Έχω όμως μια διευκρίνηση ε, να σας ζητήσω, η οποία είναι και η εξής. Τι θα γίνει με το θέμα της αναθεώρησης της στρατηγικής 2020 στους διάφορους σχηματισμούς του Συμβουλίου. Δηλαδή, Θα βασιστούμε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επόμενους μήνες. Θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Επιβεβαιώνεται τις ημερομηνίες του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλξο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα... Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ και εγώ θέλω να μιλήσω για το σχέδιο Juncker. Φαίνεται μεγαλεπίβολο και μεγαλειώδες, ίσως λόγω προπαγάνδας, 350 δις ευρώ προβάλλονται. Γίνεται λόγος για δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων απασχόλησης. Ε, μεγαλεπίβολα σχέδια. Ωστόσο, ε, βλέποντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τίθεται το εύλογο ερώτημα. Από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα, ποιε είναι οι πηγές. Ουσιαστικά θα αλλάξουμε επικεφαλίδες, θα αλλάξουμε το όνομα ε, των τίτλων και τα χρήματα που ήδη υπάρχουν σε κάποιες επικεφαλίδες θα περάσουν σε κάποιες άλλες με ένα νέο όνομα και αυτό έτσι ως εκθαύματος ε, προβάλλεται το σχέδιο Juncker. Περιμένετε τον ιδιωτικό τομέα να πολλαπλασιάσει τα δημόσια κονδύλια κατά 15 φορές. Περιμένετε τον ιδιωτικό τομέα να έχει ένα συντελεστή σε 15 προς 1. Είναι αυτό ρεαλιστικό στην έρευνα, στην παιδεία, σε όλα αυτά. Φαίνεται μεγαλειώδες, μήπως όμως είναι αυταπάτη δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι θα συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Και σύν τις άλλες, ως προς ε, ε, τη Λετωνική Προεδρία, ποιο είναι το δικό σας συγκεκριμένο καθήκον ε, κατά την εφαρμογή του σχεδίου Γιούγκερ. Ευχαριστώ κυρία Σμόλκοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι διότι στηρίζεται τη στρατηγική των μακροπεριφερειών. Έχω ένα αίτημα να υποβάλω προς εσάς και προς τη Λετωνική Προεδρία. Οι συνάδελφοί μου από την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, αλλά και από τη Σλοβακία που είναι η χώρα προέλευσής μου, και εγώ βεβαίως, προσπαθούμε ε, να τα εξετάσουμε όλα αυτά Ζητήσαμε να υπάρξει στρατηγική για τα Καρπάθια. Ζητήσαμε να οργανωθεί ακρόαση για αυτό το θέμα. Γιατί οι χώρες που είναι στα Καρπάθια έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Και αν υπήρχε τέτοια στρατηγική θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ακόμα καλύτερα και να ε, βοηθήσουμε και άλλη χώρα, την Ουκρανία σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ άλλων. Επομένως, εσείς είστε χώρα που έχετε την Προεδρία. Ζητώ να στηρίξετε την ε, πρόταση για δημιουργία μακροπεριφέρεια στον, ε, στα Καρπάθια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, αφού δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Μπόγκοβιτς. Η προσωπική μου εκτίμηση όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας. Ξεκινώντας λοιπόν την Προεδρία αυτή, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα τρομακτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Παρίσι. Εμείς όμως είμαστε μια Προεδρία η οποία έχει ένα υψηλό βαθμό ευελιξίας και καταφέραμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε προτεραιότητες ασφάλειας. Ξέρετε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν ε, ήδη δηλώσει ότι θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα στεναρά, με ιδιαίτερη πυγμή, όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως να μην απαντήσω στα ερωτήματά σας με τη σειρά που υπευλήθησαν, σας ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, όσον αφορά το σχέδιο Juncker, ή μάλλον ξεκινώντας με τη στρατηγική για τα Καρπάθια, την τελευταία ερώτηση. Εγώ υποστηρίζω την ενδεχόμενη δημιουργία μιας τέτοιας περιφερειακής στρατηγικής. Ξέρετε ότι έχουμε και μια στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής, η οποία βασίζεται στη συνεργασία των Ευρωβουλευτών της ε, Βαλτικής ε, περιοχής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και για τη δική σας την περιοχή. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί ακόμα και για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου. Νομίζω ότι η ήδη φυστάμενη ομάδα στην οποία αναφερθήκατε μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω αυτή ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία στην ε, περιοχή των Καρπαθίων, όσον αφορά τώρα τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Λοιπόν, στρατηγική Ευρώπη 2020 πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτής της στρατηγικής. Μα αυτό προφανώς εξαρτάται από τις νέες δομές οικονομικής διακυβέρνησης, εξαρτάται επίσης και από όλες τις σχετικές πολιτικές και τη χρηματοδότησή τους. Η πολιτική συνοχής προφανώς έχει συμβάλει και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων στρατηγικής Ευρώπη 2020 και η αναμενόμενη αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής προφανώς θα βελτιώσει την επίτευξη των στόχων αυτών και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και όσον αφορά τις γενικότερες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος που δραματίζει η πολιτική συνοχή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 19 Οκτωβρίου του 2014 τόνισε τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η Λετωνική Προεδρία Εκτιμά ιδιαίτερα την εργασία που έγινε από την Ιταλική Προεδρία ως προς το ζήτημα λοιπόν αυτό και θα προωθήσουμε περισσότερο μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αναθεώρηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η αναθεώρηση αυτή όμως θα πρέπει να είναι σφαιρική, θα πρέπει να χαίρει του κατάλληλου συντονισμού και θα πρέπει διάφοροι σχηματισμοί του Συμβουλίου να συμβάλλουν στην αναθεώρηση αυτή και προσβλέπω σε μια θετική συνεργασία και με εσά και ιδιαίτερα με τη δική σας την Επιτροπή. Ιδίω διότι η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η πλέον αρμόδια για την πολιτική συνοχή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στα πλαίσια επίσης της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Υποβλήθηκε και μία ακόμα ερώτηση όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να εγκρίνουμε και να εντάξουμε μάλλον στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όλες οι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον προπολογισμό για το 2015. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια διοργανική συμφωνία πριν την 1η Μαΐου του 2015, προκειμένου όλα τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην περιφερειακή πολιτική να μπορούν να ελοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Ξέρω το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και ελπίζω ότι θα καταφέρετε κι εσείς να συμβάλλετε σε αυτό επικοδομητικά προκειμένου να επιλύσουμε όλα τα κρεμή ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Αν κινηθούμε από κοινού θα καταφέρουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προγράμματα θα αρχίσουν να τρέχουν το συντομότερο δυνατό και ότι οι σχετικές επενδύσεις θα λάβουν όντως χώρα. για το επενδυτικό πακέτο Juncker. Αρχίσαμε να επεξεργαζόμαστε αυτό το σχέδιο, το σχέδιο Juncker. και θυμάμαι ένα ανέκδοτο από την ε, παιδική μου ηλικία. Ήταν λέει ένα χωριό. Ζούσαν πολλοί άνθρωποι σε αυτό το χωριό και πολλοί από αυτούς δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους ελέφαντα. Ήταν λοιπόν περίεργοι να μάθουν τι είναι αυτό το πράγμα ο ελέφαντας και ο καθένας φανταζόταν τα δικά του ποια είναι η εμφάνιση αυτού του ζώου και έτσι οι γυρεότεροι του χωριού αποφάσισαν να στείλουν μια ομάδα ανθρώπων που θα πάει να βρει έναν ελέφαντα, να τον ζωγραφίσει ώστε οι χωριανοί να ξέρουν ποια είναι η μορφή, πώς μοιάζει τελικά ένας ελέφαντας. Έφυγε αυτή η ομάδα, και μετά από λίγες εβδομάδες πράγματι βρήκαν ένα ελέφαντα, τον ζωγράφισαν και έφεραν μια ζωγραφιά στους χωριανούς. Και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση γιατί καθένας είχε τη δική του ε, ιδέα για το τι είναι ένας ελέφαντας. Πήγαν λοιπόν και κοιμήθηκαν οι χωριανοί και το πρωί η ζωγραφιά αυτή είχε διάφορες προσθήκες από διάφορους. Πήγαν και βάλαν τα δικά τους στοιχεία για να φέρουν την ε, εικόνα κοντά σε αυτό που οι ίδιοι είχαν φανταστεί. Ποιος είναι ο παραλυσμός που θέλω να κάνω. σήμερα πια. Έχουμε την ε, σύγχρονη τεχνολογία, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε ψηφιακά αρχεία και βλέπουμε ότι αυτό το σχέδιο μοιάζει με αυτόν τον ελέφαντα που σας περιέγραφα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να γίνει μια περιεκτική συζήτηση για το από, από πού θα εξευρεθούν τα χρήματα ε, θα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ποιο ποιος θα είναι ο ρόλος των διαφόρων παικτών. Αλλά σε πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, να καταλάβουμε τι θέλουν τα κράτη-μέλη από μας και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό ε, σχέδιο. Για μένα λοιπόν η μεγαλύτερη ε, πρόκληση είναι το σχέδιο αυτό από ελέφαντας να μην καταστεί ξαφνικά ένα τέρας, ένα θηρίο, αλλά να εξυπηρετήσει τους στόχους για τους οποίους εκπονήθηκε. Γνωρίζω ότι οι συζητήσεις θα είναι πολύ δύσκολες και εσείς εδώ εντός αυτής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου έχετε τις διαφωνίες σας. Υπήρχαν πάρα πολλές προσδοκίες στις ακροάσεις των Επιτρόπων και στο Συμβούλιο, αλλά θα καταβάλει ο καθένας τις δικές του προσπάθειες για να στεφτεί με επιτυχία το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που θα γίνει στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ τον Φεβράριο ή τον Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει συμφωνία ότι πρόκειται για ένα ε, στατικού χαρακτήρα επενδυτικό ε, πακέτο δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις αλλά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα ε, τις υπάρχουσες επενδύσεις και τα χρήματα θα εξαιρεθούν εν μέρη και από ε, ιδιωτικούς πόρους. Τα κράτη-μέλη θα παρουσιάσουν επενδυτικά σχέδια και μάλιστα τα, αυτά που έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν και τα 350 ε, δισεκατομμύρια και το μεγαλύτερο μέρος ε, των χρημάτων θα προέλθει από ιδιωτικούς πόρους, από ιδιώτες επενδυτές. που θα υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση των ε, έργων ε, ε, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Οι διαγωνισμοί θα είναι ανοιχτοί. Προς το παρόν δεν έχουν οριστεί προθεσμίες για την υποβολή σχεδίων έργων και βεβαίως ενθαρρύνονται και οι ιδιώτες επενδυτές για συμμετοχή. Και στόχος δεν είναι μόνο να εξευρεθούν χρήματα για συγκεκριμένα έργα και δράσεις, αλλά ε, στόχος μας είναι να υπάρξει και μια αναδιαμόρφωση της αγοράς, να ενισχυθεί, να γίνει πιο ανθεκτική, να γίνει ε, μια απολοποίηση της νομοθεσίας και θα ήθελα να πω ότι η Προεδρία δίνει ε, μεγάλη σημασία σε δύο στοιχεία. Αφενός στο ψηφιακό θεματολόγιο θα προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε τις ε, συζητήσεις στον τομέα αυτό και η ενεργειακή αγορά, η αγορά ενέργειας που νομίζω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί στο τέλος αυτό το σχέδιο, το επενδυτικό σχέδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπω είπα, ε, περιμένουμε τις ε, συζητήσεις των κρατών μελών και το ΕΚΟΦΗΝ του Μαρτίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μάλλον θα ξανασυναντηθούμε και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Με, αφού ληφθούν οι αποφάσεις στο ΕΚΟΦΗΝ και αφού ε, καταφέρουμε και εμείς να ε, καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και εμείς θα συζητήσουμε για αυτό το επενδυτικό σχέδιο εδώ στην Επιτροπή μας και αν δεν υπάρχουν ε, άλλες ερωτήσεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας, για την παρουσίαση σας ε, για τις προτεραιότητες της Λετρονικής Προεδρίας ε, όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή. Σας ε, ε, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας και δεσμευόμαστε ότι θα υποστηρίξουμε στο μέτρο του δυνατού ως Επιτροπή. Και σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε στενά το έργο της Προεδρίας σας. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόσκληση που απευθύνατε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Προσβλέπω στην συνεργασία μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Θα τα ξαναπονούμε σύντομα. Συνάδελφοι, θα γίνει ψηφοφορία στις 10 και Να αποχαιρετήσω τους ε, καλεσμένους μας και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Okay, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε σήμερα το κείμενο για την απαλλαγή του 2013, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκέλος που αφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή για τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού, καταρτίζει αυτή τη στιγμή την έκθεσή της χορηγώντας απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2013. Η Επιτροπή ζήτησε ε, τις ε, άλλες επιτροπές να στείλουν τις γνωμοδοτήσεις τους μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Οι συντονιστές της Ρέτζη ε, όρισαν την πρόεδρο ως... Ε, συντάκτη της γνωμοδότησης. Ε, καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν η 11, η Δεκεμβρίου. Είχαμε 38 τροπολογίες που υποβλήθηκαν και μετά από διαβούλευση με τους σκιώδεις εισηγητές και τους συμβούλους πρότεινα 8 συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής μας για τη συνεισφορά τους, για τις, για τις τροπολογίες τους και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους συζητήσαμε το ε, κείμενο ε, προς, που θα είναι το αντικείμενο του συμβιβασμού. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στη ψηφοφορία. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας, έτσι δεν είναι? και μπορούμε να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά εάν χρειαστεί, όπου δει. Ξεκινούμε λοιπόν με τη συμβιβαστική τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 30 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τέλος, ε, η τελική ψηφοφορία επί του κειμένου θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, μία ψήφος κατά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι καταχωρήθηκε ε, η ψήφος μου, γιατί έχω χάσει την κάρτα ψηφοφορίας μου. Ναι, ευχαριστούμε. Η ψήφο σας είναι υπέρ, άρα έχουμε 34 ψήφους υπέρ και μία κατά. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά. Καλώς. Πρέπει να εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Τις έχετε. Έτσι δεν είναι. Εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Ναι τι εγκρίνουμε. Υπάρχει κάτι υπό τα διάφορα. Θέλετε κάτι άλλο να θέσετε ως θέμα. Όχι. Να σας υπενθυμίσω ότι θα συνεδριάσουμε την 5η 26 Φεβρουαρίου ξανά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6.30 το βράδυ. Να ευχαριστήσω τους δερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Λέει Πρόεδρος, ευχαριστούμε και εμείς. Κυρίσω το πέρα στη συνεδρία σας.